δεν υπάρχουν ενστάσεις ε, στους διορισμούς ε, αυτούς, θα θεωρηθούν εγκεκριμένοι. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ μας διαβιβάσε διορθωτικό για κείμενο του Κοινοβουλίου και βάσει του άρθρου 231 θεωρείται εγκεκριμένο αυτό το διορθωτικό. Εάν εντός 24 ώρων δεν έχουμε ένσταση από πολιτική ομάδα ή από τουλάχιστον 40 βουλευτές, ε, θα ψηφιστεί το κείμενο, θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος ε, θα σας ε, δημοσιευθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Την ε, Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω δύο νομοθετικά